πολιτική οικονομικού συντονισμού και τις προτεραιότητες για το 2014. Η έκθεση υποβλήθηκε από τον Νίλ Στόρβαλς. Ε, υποβλήθηκαν 28 τροπολογίες, ενώ ο εισηγητής προτείνει 4 συμβαστικές τροπολογίες. Θα δώσω το λόγο στον Νίλ Στόρβαλς για να μας πει ποια είναι η αποψή του για τις συμβασικές του απολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα περισσότερα αναφέρθηκαν ήδη νωρίτερα. Κάποιες μικρές διορθώσεις στο συμβιβαστικό κείμενο είναι τα εξής μια προφορική τροφολογία, αν κατάλαβα καλά, θα υπάρξει από τους σοσιαλιστές. Πάντως ο κατάλογος της είναι παρκώς σαφής. Ευχαριστώ. Très Ωραία. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Τροπολογία 1. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Δεν υπάρχει κανείς κατά, ούτε αποχές. Τροπολογία 2. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κάτω τα χέρια. Κατά. Ουδής. Αποχή καμία επίσης. Συμβαστική τοπολογία 1. Για την παράγραφο 2. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αντίθετη. Δύο. Αποχές. Καμία. Μια διευκρινιστική τροπολογία υπαριθμών τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη διευκρινιστική τροπολογία Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 για την παράγραφο 3 βάσει των τροπολογιών 6 και 7 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. 2. Αποχές. Καμία. Το συμβιβαστική 3 βάσει των τροπολογιών 8, 9 και 10 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Δύο. Αποχές. Παράγραφος 5. Τροπολογία 11. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. αποχές, πέντε αποχές. Απορρίπτεται. Amendement numéro 12. απολογία 12. Και εδώ η εισηγητής είναι κατά. Όσοι είναι υπέρ, να σηκώσουν το χέρι τους. Ευχαριστώ. Κατά. Κατεβάστε τα χέρια σας. Αποχή. Δεν υπάρχει καμία αποχή. Απορρίπτεται η τροπολογία. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Βάση των τροπολογιών 13-14-15 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρει, κατά. Αποχέ. Καμία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Η τροπολογία 16. Ο εισηγητή είναι κατά. Υπέρ τις 16. Κατεβάστε τα χέρια σας. Αντίθετη. Ευχαριστώ. Ποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά καλύτερα να γίνει ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 κατά 13. Τι θέλει να ξαναψηφίσουμε. Ξαναψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ξανά. Ξαναψηφίζουμε λέω. Ah bon, pardon. Oui. Alors on doit reprendre. Θα ξαναρχίσουμε. C'est bon. <laughs> Très bien. Le scrutin est clos. ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 14 κατά, 3 αποχές. Παράγραφος 8. Το Τροπολογία 19. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Είναι κατά, συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Αντίθετη αποχές απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 20. Και εδώ η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Με θετική γνώμη του εισηγητή. Υπέρ. Κατά ούτε αποχή εγκρίνεται η τροπολογία. Παράγραφος 9, τροπολογία 23. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, 25 τροπολογία ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Έχω αμφιβολίες για το αποτέλεσμα. Άρα θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 18 υπέρ, 15 κατά. Παράγραφος 10α. Προσθήκη. Τροπολογία 26. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. 27. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ της 27. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά να το κάνουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 28. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 19 κατά, 14 υπέρ, 3 αποχές. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τοποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Πέρας ψηφοφορίας. Το κείμενο όπως τοποποιήθηκε εγκρίνεται. 28 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές. Nous allons maintenant procéder au vote des quelques 1500. Τώρα θα ψηφίσουμε γύρω στις 1500 τροπολογίες των επιτροπών, των ομάδων και των λοιπόν συναδέλφων για την θέση του Συμβουλίου ως προς το σχέδιο προϋπολογισμού 2015. Σημειώστε ότι θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα 7 Οκτωβρίου το ψήφισμα που θα συνοδεύσει τις τροπολογίες όταν περάσουν στην Ολομέλεια κάτι που προγραμματίζεται για τις 22 Οκτωβρίου. Συμφωνήσαμε να ψηφίσουμε με την εξή σειρά. Θα εξετάσουμε πρώτα τις τροπολογίες για τις πιστώσεις για τις υπηρεσίες και οργανισμούς. Κατόπιν την ε, στήλη, την κατηγορία 5. Μετά την κατηγορία 1β, την κατηγορία 2, 3 και ίσως στις 6.30 να τελειώσουμε. Κάτι που σημαίνει ότι αύριο θα εξετάσουμε τις τροπολογίες για την κατηγορία 1α και την κατηγορία 4, τα ειδικά μέσα και τις πιστώσεις για τα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, τις άλλες, τα άλλα τμήματα και τις πληρωμές εν τέλει. Κάθε κατηγορία ψηφοφορίας ακολουθεί τον γενικό κανόνα που είναι ως εξής. Οι προτα... συμβαστικές προτάσεις του εισηγητή θα τίθενται σε ψηφοφορία πρώτα. Υπό τη μορφή ομάδων, πακέτων, μπλοκ, Κατόπιν, αν χρειαστεί, θα ακολουθήσει ψηφοφορία για τις ατομικές τροπολογίες που δεν καλύπτονται από τα συμβαστικά κείμενα ή για τις οποίες θα ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία από μία ομάδα μέσα στις ε, προθεσμίες που έχουν τεθεί. Σε περίπτωση που εγκριθεί μία χωριστή ψηφοφορία θα υπερισχύσει τη συμβαστικη προτάσεως. Κατόπιν θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες για τις παρατηρήσεις και τα αποθεματικά. Τα μέλη της Επιτροπής παρακαλούνται να κοιτάξετε τον κατάλογο ψηφοφορίας που έχει γίνει για κάθε ομάδα, τα παρατήματα που περιέχουν το πακέτο συμβαστικών προτάσεων και το κείμενο 4 που έχει το σύνολο των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Ευχαριστώ τους εισηγητές μας και γενική εισηγήτρια και εισηγήτρια για τα άλλα τμήματα που ετοίμασαν την συζήτηση που θα μας επιτρέψει ίσως να κερδίσουμε και χρόνο και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την εξέταση και την ψηφοφορία. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, το γενικό εισηγητή κυρίω, ίσως η κυρία Καλίνιο, Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού στην Επιτροπή, θέλει να μας παρουσιάσει την άποψή της και να μας προετοιμάσει για την εξέταση των τροπολογιών. Έχετε το λόγο. Με ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να σας απευθυνθώ να σα απευθύνω το λόγο για τη σημαντική αυτή ψηφοφορία που θα ψηφίσουμε για την διαδικασία προπολογισμού του 2015 στι πέρασμένε συναντήσει και στου τρομερεί διαλόγου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προτάσεις για τον προπολογισμό του 2015 και να ε, εκφράσει την απόψη της για την ανάγνωση του Συμβουλίου. Σήμερα λοιπόν διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι οι πολυάριθμες τροπολογίες των Ευρωβουλευτών από πλευρά των ειδικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό θέλουν να επανέλθουμε στο, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, δεσμεύσει πληρωμών στο σχέδιο προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει ε, ε, πληρωμών, σε ό,τι αφορά το 1α και το 4, θα επανέλθουμε σε ό,τι αφορά τι ε, προτεραιότητέ μα για να ενισχύσουμε την απασχόληση διεθνή, στο διεθνέ προσκήνιο. Δεν χρειάζεται να σα υπενθυμίσω ότι ο προπολογισμό αφορά τι επενδύσει, άρα δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανάπτυξη και θέση απασχόληση και εκ παραλίλου να περικόπτουμε τι δαπάνε τους τίτλους εκείνους ακριβώς που συμβάλλουν ε, ως επιτοπλίστων στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Οι επενδύσεις λοιπόν θα πατώσουν καρπούς αν υπάρχουν οι ανάλογες πληρωμές το 2015 και τα επόμενα χρόνια. Άρα, χαίρομαι που βλέπω ότι μία σειρά, μεγάλη σειρά τροπολογιών προτείνουν να επανέλθουν τα επίπεδα πληρωμών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό διορθώνει ουσιαστικά την μείωση κατά 2 δισεκατομμύρια την οποία έχει προτείνει το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι μια σειρά τροπολογιών που έχουν προταθεί για να αυξηθούν οι δεσμεύσει πληρωμών πέρα από τι ε, προτασίες ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπερνούν το ε, ανώφλι του, του δημοσιονομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την περίοδο του 2013. Κατανοώ ότι απότερο στόχο είναι προφανώ να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του backload, αλλά ότι αυτά τα προβλήματα πληρωμών θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστικό τρόπο το 2015. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη αν ε, εγκριθεί το, αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 4,7 σε μέχρι τα 30 δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2015 θα είναι ρεαλιστική και σόφρον ε, η προσέγγιση για να αναπτυχθούν τα προγράμματα επενδύσεων που είχαμε συμφωνήσει μέχρι το 2020. Γιατί σκοπός μας είναι εφαρμοστεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θεωρούμε ότι η πρότασή μας αποτελεί ένα ρεαλιστικό τρόπο για να το πετύχουμε αυτό. Ελπίζουμε ότι οι επικοδομητικέ συζητήσει τη περασμένη εβδομάδα μεταξύ των θεσμικών οργάνων σα επέτρεψαν να σχηματίσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα και εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για την οργάνωση της τη αυτή. Κάποιε σύντομε παρατηρήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια που προτείνει να επανέλθουν τα επίπεδα δεσμεύσεων πληρωμών σε ό,τι αφορά τη διοίκηση και την διοικητική υποστήριξη που χρειάζονται για την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω στο σημείο αυτό τον περιορισμό που έχει αυτοεπιβληθεί, την αυτολογορικήσια που έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η κοινή στόχη της πιο αποτελεσματικής ε, διοίκησης έχουν μπει και στους στόχους σε ό,τι αφορά τη μείωση κατά 5% τα επόμενα 5 χρόνια των εξόδων για το προσωπικό. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε με την πρότασή μας. Προτήσαμε συνολική μείωση 1% σε ό,τι αφορά τα σχέδια εγκαθίδρυσης όλων των θεσμικών οργάνων και κυρίως των αποκεντρωμένων οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των νέων οργανισμών που ε, καλούνται να εκτελέσουν νέα καθήκοντα. Και σημειώνουμε ότι μία σειρά τροπολογιών που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή προτείνουν να αυξηθούν ε, τα έξοδα και οι δαπάνες κάποιων αποκεντρωμένων οργανισμών κατά 200 20 ε, μέλη προσωπικού. Αυτό θα σήμαινε αύξηση 2,5% πάνω από το... τα επίπεδα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία δεύτερη παρατηρήση, την οποία θα ήθελα να κάνω, έχει να κάνει με την πρόταση της ε, εισηγήτριας των εισηγητριών να, να μεταφερθούν δαπάνες από το τμήμα για την υπηρετησία εξωτερική δράση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά το, το κεφάλαιο, το, το τμήμα, τη γραμμή 5. Αυτό θα σημαίνει μια απλοποίηση. Και υπάρχει μια πρόταση τη κυρία Χολμάιερ να μεταφερθούν δαπάνες που έχουν να κάνουν με τα κοινά έξοδα στον προϋπολογισμό της εξωτερικής υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Καταλαβαίνω τους λόγους ε, που γίνεται αυτή η πρόταση τροπολογίας για λόγους απλούστευσης προφανώς, αλλά εκ παραλλήλου είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι θα καταργούσαμε τη σύνδεση μεταξύ του, της και του υποστηριζόμενου προγράμματος. προγράμματος. θα πρέπει να είναι ουδέτερη από πλευρά δημοσιονομική αυτή η αλλαγή. Και τέλο, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά προγράμματα και τι προσπαραβασκευτικέ δράσει, υπάρχουν κάποιε νέε ιδέε σε ό,τι αφορά την πολιτική. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να σα βοηθήσουμε να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τι τελικέ προτάσει που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτό. Τέλο, μία σειρά τροπολογιών που προτείνονται Προτείνω το σχηματισμό ενός ε, αποθεματικού το οποίο θα απελευθερώνεται μόνο υπό κάποιους όρους. Θα ήθελα να γίνει μια πλήρης αξιολόγηση από την Επιτροπή, από την Επιτροπή σας σε ό,τι αφορά το κατά πόσον είναι πραγματικά σωστή αυτή η όρη, αυτές οι συνθέκεις. Κατά πόσον υπάρχει άμεση σύνδεση, κατά πόσον υπάρχει και διακυβεύεται η ανεξαρτησία των θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα ιδιαίτερως να αναφερθώ στο αποθεματικό που έχει να κάνει με την ανεξαρτησία και την ιδιωτερότητα των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αδιαφάνεια, μια έλλειψη ισορροπίας στη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά το σχηματισμό και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων και το Κοινοβούλιο έχει κάνει προτάσεις σε ό,τι αφορά την αποζημίωσή τους και σε ό,τι αφορά το σχετικό μητρό που υπάρχει. Θα εξετάσουμε και τη σχετική έκθεση του διαμεσολαβητή, θα συνεργαστούμε με τον διαμεσολαβητή, αλλά δεν συμφωνούμε να υπάρχει τέτοια πρόοδος στον τομέα αυτών. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο όργανο για να πετύχουμε την καλύτερη οργάνωση των ομάδων εμπειρογνωμόνων μας. Μία σειρά τροπολογιών προτείνουν να αλλάξουν οι στόχοι κάποιων προγραμμάτων ε, και να μπουν ε, κάποιες νέες ε, επικεφαλίδες. Θέλουμε λοιπόν να σεβαστούν τους όρους των προγραμμάτων τα οποία το οποίο είναι κάτι το οποίο θα, σίγουρα θα σας, ε, με το οποίο θα συμφωνήσετε σίγουρα. Και να πω ότι προσβλέπουμε στην ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα σήμερα και θα πρέπει να σας ε, παρέχουμε και μια επιστολή ε, εφαρμοσιμότητας για να δούμε κατά πόσον οι προτάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και πώς μπορούν να εφαρμοστούν με το βέλτιστο πνευματικό τρόπο. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, η, Ευρωπαϊ... Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις που σας έκανα και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Σίγουρα θα προχωρήσουμε. Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των τροπολογιών, η Γενική Συγγήτρια θέλει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτον, μια και μίλησε η Επιτροπή, να την ευχαριστήσω για την δουλειά που έκανε και για την υποστήριξη που μας έδωσε στην προετοιμασία του σχεδίου προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και τις πολιτικές ομάδες προφανώς, τους συντονιστές, για την υπομονή που έχουν δείξει. Ποτέ δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε πάνω από 1.400 τροπολογίε και να βρούμε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλε τι ομάδε. Θέλω να καταστήσω σαφέ πάντω ότι ο στόχο με την πρόταση που θα ψηφίσουμε σήμερα και αύριο κατά βάση έχει στόχο να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που εμείς ως Ευρωβουλευτές ε, υιοθετήσαμε, αλλά και το υπογραμμίζω αυτό με τις δεσμεύσει που και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει την κάθε φορά που, κάθε φορά που συναντιέται. Να χρησιμοποιήσω λοιπόν όσο περισσότερο και όσο καλύτερα γίνεται τους ε, πόρους που υπάρχουν στα προγράμματα που θεωρούμε ότι είναι πολιτικές προτεραιότητες για μας. Την ίδια λογική έχουμε και στις πληρωμές. Η μόνη πρόταση του Κοινοβουλίου είναι να πληρώνουμε αυτά που οφείλουμε και μπορώ να καταλάβω απόλυτο ότι η Κομισιόν ε, υποβάλλει μια προσεκτική πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά εμείς ως Ευρωβουλευτές και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ε, κλάδος της Δημοσιονομικής Αρχής, θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι οι πρώτες προϋπολογισμού μας παρέχει επαρκή, επαρκή κονδύλια για να πληρώσουμε αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε το 2015 και επιπλέον κονδύλια για να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτά που δεν πληρώσαμε τα προηγούμενα έτη. Γι' αυτό η πρόταση πάει στις πληρωμές παραπέρα από την προσεκτική ανάγνωση που ανέφερε η Επιτροπή. Ευχαριστώ εκ νέου όλους όσοι μετέσχουν στην ε, διαμόρφωση της κοινή αυτής θέσης του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι οι ψηφοφορίες δεν θα είναι πολύ περίπλοκες. Μία τεχνική λεπτομέρεια. Αναφέρθηκε και η Επιτροπή, το συζήτησα και με την εισηγήτρια για τους Σαγετάλα του χόλμα. Χολμάγερ, υπάρχει ένα σημείο που ανήκει στους δύο προϋπολογισμούς, και το τρία και τα άλλα τμήματα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και Κομισιόν, τις οποίες δεν διαθέτουμε ούτε τις λεπτομέρειες όλες, ούτε την προβληματική που καλύπτει. Για να αποφύγουμε λοιπόν κάτι εσφαλμένο σήμερα ή να ψηφίσουμε κάτι που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη δουλειά της Επιτροπής στο μέλλον, θα καθυστερήσουμε την ψηφοφορία αυτή μέχρι αύριο και ή δυνατόν και μέχρι την Ολομέλεια. Όταν μέχρι ότου υπάρξει σαφές, καταστεί σαφές πώς είναι η συμφωνία και ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι τεχνικά μπορεί να γίνει και δεν θα ήθελα να ψηφίσουμε κάτι που δεν μεταφέρει ακριβώς τη συμφωνία που έχουν συνάψει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ και ευχαριστώ εκ νέου για την βαριά δουλειά που αναλάβατε και που μας επιτρέπει σήμερα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με ξεκάθαρα τα θέματα. Κύριε Χολμάγερ, και εσάς ε, σας αφορά το θέμα των αποθεματικών για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε να πείτε κάτι? Καταρχάς να πούμε ότι ξέρουμε πλέον ακριβώς τι ψηφίζουμε. Έχουμε τον κατάλογο όλοι μας μπροστά μας το κατάλογο ψηφοφορία και ο φόβο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Συμβούλιο ενδεχομένω θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να κάνει περικοπέ, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει διαφανεί τέτοια τάση. Αλλά σίγουρα αυτό θα το κοιτάξουμε τελευταία στιγμή και θα ήθελα να προτείνω το εξή αύριο να ψηφίσουμε. Μέχρι τότε θα έχουμε και τις δηλώσεις του, του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον δεύτερο προπολογισμό. Είναι σαφείς οι γραμμές δημοσιονομικές, είναι σαφείς οι θέσεις σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν το Συμβούλιο δηλώσει ότι δέχεται τον ουδέτερο αυτοπροπολογισμό προπολογισμό, θα διευκρινιστεί η κατάσταση και θα ψηφίσουμε αύριο. Très bien, je vous remercie. En écho propos de... Ωραία. Να τονίσω και εγώ, όπως είπε και η Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής, ότι η συνάντηση της 24 η Σεπτεμβρίου ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, αν και μας απογοήτευσαν οι απαντήσεις του Υπουργού, που δεν αμφισβήτησε το ποσό του χρέους, αλλά η εξέταση του σχεδίου υπολογισμού 15 θα ήταν απλούστερο αν είχαμε μια σαφή εικόνα ε, πληρωμής του, των χρεών, το ώστε να μην χρειαστεί να κινητοποιούμε όλα τα μέσα που μας διαθέτει ο υπερπολογισμός για να ξεκινήσουμε να σταθεροποιούμε την κατάσταση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την εξέταση των τροπολογιών και να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Ηλεκτρονικά θα γίνονται οι ψηφοφορίες, άρα ετοιμάστε τις κάρτες σας. Το έχετε όμως, γιατί ήδη ψηφίσαμε προηγουμένως, ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ξεκινούμε με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς. Nous avons Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει ψηφοφορία όλων μαζί των ε, τροπολογιών όσον αφορά τι ε, πιστώσει ακριβώ όπω έχουν εγγραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ όσον αφορά την έγκριση όλων μαζί αυτών των τροπολογιών. Έναρξη ψηφοφορία. Pardon ναι. Ηλεκτρονικά, ναι, λέει ο πρόεδρο. Ε, Γενική Συγκέντρια. κύριε Πρόεδρε, σας προτείνω να ψηφίσουμε με ανάταση τη χειρό ω συνήθω, γιατί υπάρχουν και κάποιες ψηφοφορίες που μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, κάποιες. Καλά, αν δεν υπάρχουν ε, αμφισβητήσει όσον αφορά το πιο πώς διαμορφώνεται η πλειοψηφία, καλά, κερδίζουμε χρόνο. Και τώρα, όσον αφορά την επαναφορά των πιστώσεων. Σηκώστε χέρια, σας ευχαριστώ. Κατά. Πέντε κατά. Άρα, εγκρίνεται. Πάμε τώρα σε μια δεύτερη ομάδα τροπολογιών που προβλέπουν για κάποιες πιστώσεις πέραν των όσων είχαν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιοι είναι Υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Πέντε κατά. Επομένως συγκρίνεται αυτή η ομάδα τροπολογιών. Και τώρα. Στο οργανόγραμμα, αλλά όσον αφορά την δημιουργία θέσεων, θα ψηφίσουμε όλες μαζί αυτές τις ε, τροπολογίες αφορούν τη δημιουργία 184 θέσεων για αυτές τις περισσότερες οργανισμούς. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Είναι κατά. Αποχές. Δεν έχουμε αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογική τώρα. Στις ε, παρατηρήσεις, υποσημειώσεις. 6665. Pour. Είναι υπέρ ποιοι είναι υπέρ, κατά, κατά, τρεις είναι κατά αποχές. Εγκρίνεται αυτή η τροπολογία. 82-72 Εδώ είναι κατά η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ για αυτές τις τροπολογίες. <laughs> Κατά, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ, αποχές. Δύο αποχές και αυτή απορρίπτεται. 12.03.02 Υπέρ η συγγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. 5 είναι κατά, εγκρίνεται. Είναι το, το κονδύλιο 12.03.03, είναι υπέρ εισηγήτρια, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τέσσερις είναι κατά, αποχές. Μία αποχή. Πάμε για το... 12.03.04. Ε, υπέρ εισηγήτρια, ποιοι είναι υπέρ. Σε ευχαριστώ. Κατά πέντε είναι κατά, αποχές δεν έχουμε, εγκρίνεται. Όσον αφορά τώρα τα αποθεματικά, 18.02.03 είναι το κονδύλιο. 61.01 ε, είναι υπέρ εισηγήτρια, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, τρεις είναι κατά, όχι τέσσερις λέει ο πρόεδρος, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα 79-17. Ποιοι είναι κατά εισηγήτρια, ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Απορρίπτεται. Ταυτόσημη. 42-01, άρα το ίδιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε για οργανισμούς και υπηρεσίες. Και τώρα, προχωρούμε. 3. Στο τρίτο τμήμα. Διοικητικές δαπάνες. premier amendement. Πρώτη τροπολογία. À la section 3. Η πρώτη του Εδώ ο σκοπό είναι να αποκατασταθούν κάποια κονδύλια τα οποία είχαν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπέρ. Κατά. Six avis contraires. L'amendement. Έξι είναι κατά, που μόνο συγκρίνεται. Τρίτο τμήμα κεφάλαιο παριθμών 5. Επαναφορά των πιστώσεων. Και εδώ θα πιστώσουμε, θα ψηφίσουμε όλες μαζί τις ε, τροπολογίες υπέρ η συγγήτρια, ποιοι είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Κατά. Έξι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μεταφορά πιστώσεων δεν θα ψηφίσουμε τώρα γιατί η Γενική Εισηγήτρια ήθελε να επιφυλαχθούμε όσον αφορά την ψήφιση. 0401, 0402 το κονδύλιο. Σε αυτό ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουμε αποχές. Απορρίπτονται. Η επόμενη τώρα είναι κατά εισηγήτρια, ένα σημείο υπέρ, ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Ίδιο. 79-56. Είναι υπέρ η συγκίτρια. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. que nous pourrions faire un vote. Νομίζω τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε όλε μαζί τις ε, τροπολογίες 84 και 83 όλες ε, ε, υπέρ εισηγήτρια ποιοι είναι υπέρ κανείς πώς pardonnez-moi. Les amendements 84 84-82. Είναι κατά εισηγήτρια. Και 84-85. 84-84. 84-83. Κατά εισηγήτρια. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε αυτές όλες μαζί. Συμφωνείτε. Αφού θα ψήσουμε όλες μαζί, πέστε μας ποιοι είναι υπέρ. Κανείς. Α, τέσσερις είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ευχαριστώ τελικά στα χέρια σας. Άρα, αυτές οι τέσσερις τροπολογίες απορρίπτονται. Από κάτω. 03-01-03. Είναι κατά εισηγήτρια, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 41-78. Κατά η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτωται. Απορρίπτονται. 41-79. Είναι υπέρ. Η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41-80. Κατά. Η που πηγαινε πήγαινε υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43-14. Κατά. Η Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 31-01-07-01 43-15 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42-92 κατά εξηγείται υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 31-01-08-01-43-16 Υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται 41-67 Ποιοι είναι υπέρ κατά απορρίπτεται στις παρατηρήσεις σχόλια 25.01.12 είναι το κονδύλιο και είναι η τροπολογία 41.22 κατά ισχύς υπέρ κατά απορρίπτονται 43-73 είναι κατά η συγκίτρια ποιοι είναι υπέρ κατά η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται 19-18 31-01-07-01 η τροπολογία 42-92 κατά η συγκίτρια ποιοι είναι κατά αποχές Τώρα για τα αποθεματικά. Για το κονδύλιο 24-01-07. Κατά εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται η τροπολογία. Όχι. Απορρίπτεται, λέει ο Πρόεδρος. 16, 19 και 2 εποχές. Κονδύλιο 0102 1102 4368 Υπέρ συγκεκριά Υπέρ Κατά Τρεις κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Το 869, επομένως, το δεν ψηφίζεται. Καλύπτεται. Ολοκληρώσαμε τώρα όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες για το τρίτο τμήμα. Και Πάμε παρακάτω. Πάμε στο τμήμα 1β. Εκεί έχουμε και κάποιες καταδιέρεσεις ψηφορίες χωριστές. την 040601 fad η εισηγήτρια προτείνει την τροπολογία 7548 για την συμπερίληψη κονδυλίων πιστώσεως άνω του προσχεδίου προσυπολογισμού. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. 2, 3, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η επόμενη τοπολογία λόγω της ψηφοφόρια που κάναμε τώρα. 04-04-01. Ίδια διατύπωση, ίδια, ίδιο σχόλιο. une minute, vous. Μισό λεπτό. Voilà, pardonnez-moi. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μπορεί να κάνουμε ψηφοφορία ομαδικά για τις 4307 79-31 ε, και 79-37 αν συμφωνούμε τρεις τροπολογίες λοιπόν ποιοι είναι υπέρ των τριών αυτών τροπολογιών η συγγήτρια είναι κατά τέσσερις τροπολογίες διορθώνει ο πρόεδρος 43-07 43-0-0, 79 79-31 και 79-37 ποιοι είναι υπέρ να σηκώσουν τα χέρια τους Ευχαριστώ. Κατεβάστε τα χέρια σας. Ποιοι είναι κατά των τεσσάρων τροπολογιών υπέρ. Ε, αποχές Δύο. Οι το, τέσσερις αυτές τροπολογίες απορρίπτονται. Αποθεματικά. 13.04.60. Τροπολογία 45.69. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ της τροπολογίας Ευχαριστώ. Κατεβάστε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρατηρήσεις. Σχόλια, συγγνώμη. Θα ψηφίσουμε ομαδικά για τις 8071, 8070, 8073, 8072, 8067, 8074, 8068 και 8075. Η συγγήτρια είναι κατά όλων των τροπολογιών. Ψηφίζουμε ομού. Υπέρ των τροπολογιών. Κανείς δεν σήκωσε χέρι του. Κατά. Απορρίπτονται. Σχόλια. H1β. 0402 γραμμή. Πρώτη τροπολογία 65-53. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 83-41 είναι ταυτόσχρονη. Άρα εγκρίνεται και αυτή. 79-31 ε, η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατεβάστε τα χέρια σας κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω. 40-72. ζητήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 79-31 ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19-14, τέσσερις εποχές. Η τροπολογία 40-72, η εισηγήτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. 3 κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Τρεις εποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. ...62-54 στην γραμμή 06 Η συγγυητρία είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79-36 τροπολογία. Η συγκιτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. 42-20 είναι ίδια. Τροπολογία 43-41. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Τρεις. Εγκρίνεται. 02 01 ε, γραμμή, το υπολογία 66-80, η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 8034 στη γραμμή 130363 η συγγήτρια είναι κατά υπέρ ευχαριστώ κατά ευχαριστώ αποχές καμία απορρίπτεται κλείσαμε και με τις ψηφοφορίες για την κατηγορία 1β. Κατηγορία 2. Θα δώσω το λόγο στη Γενική Συγγήτρια για τις πληροφορίες στην κατηγορία 2. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι υπάρχει μια μικρή αλλαγή στον κατάλογο ψηφοφοριών. Μετά τη συνάντηση των συντονιστών, όπου τελικά επέλθε συμφωνία, θα βάλουμε 5 εκατομμύρια ευρώ στη γραμμή 110660 η τροπολογία αυτή είναι απόδειξη της υποστήριξης προς τους αλληλείς που μπορεί να επηρεαστούν από την, το εμπάργο από τη Ρωσία των γεωργικών και των αλευτικών προϊόντων. Για τα γεωργικά είχαμε μια συμφωνία 30 εκατομμύρια ευρώ που ήταν μέσα στον κατάλογο. Τώρα υπάρχει μια συμφωνία για 5 εκατομμύρια για τις ζημιές στην Αλία. Θα αποτελούσε τμήμα του δεύτερου υπομπλοκ και θα το ψηφίσουμε σαν χωριστή γραμμή. Όταν ψηφίσουμε δηλαδή το μπλοκ των γραμμών που ξεπερνούν την πρόταση της, που υπερβαίνουν την πρόταση της Επιτροπής, θα συμπεριληφθεί και αυτή η αλλαγή. Δεν θα χρειαστεί να ψηφιστεί χωριστά. 5 εκατομμύρια ευρώ για τους αλληλείς που πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο. και μετά λένε ότι κάνουμε περικοπές συνεχώς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρώτη υποομάδα αποκατάσταση των πιστώσεων που είχαν προβλεφθεί αρχικά από την Επιτροπή πίνακας 3 του παρατήματος. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας. Κατά. Έξι κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. Δεύτερη υποομάδα. Η υπέρβαση της γραμμής ε, που είχε θέσει, των γραμμών που είχε θέσει η Επιτροπή, των ορίων που είχε θέσει η Επιτροπή, όπως επίσης το βλέπετε στο παράτημα του πίνακα 4. Η εισηγήτρια είναι υπέρ και εδώ. Ποιοι είναι υπέρ, Ευχαριστώ. Ψήφι κατά. 6. Και αυτή η τοπολογία εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στις τις τοπολογίες που δεν καλύπτονται από τους συμβασμούς. 02 0502-03, τροπολογία 621 και 872. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Δύο υπερψήφισαν. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται η τροπολογια 05-02-10-01 01 γραμμή του προπολογισμού. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας που προτείνει χωριστή ψηφοφορία για 30 εκατομμύρια υπέρβασης του σχεδίου προπολογισμού που είχε καταθέσει η Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής. Ναι, ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Ευχαριστώ. αποχέ. Τρεις. Τέσσερις. Εγκρίνεται. Η 244 Η 2.42 έχει καταπέσει, συγγνώμη. 05.02.11.99 γραμμή. Τροπολογία 41.55. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Τρεις. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 0502-1301, 622 και 870 τροπολογίες. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Γραμμή 0502-1505, τροπολογία 623 και 869 και εδώ είναι κατά εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καμία. Η τροπολογία απορρίπτεται. Γραμμή 0503-0101. Τροπολογία 627. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 05-03-01-02. 624 τροπολογία. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Τρει ψήφοι κατά. Τρει ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται η τροπολογία. Σχόλια γραμμη 05-02, 05-99. Τροπολογία 53-45. Ο εισηγητής είναι κατά. Η εισηγήτρια, συγγνώμη, είναι κατά. Υπέρ. «53-45 τροπολογία. είχε τροποποιηθεί η προηγούμενη τροπολογία. Για την 5345 ρωτώ, ποιοι είναι υπέρ, η συγγήτρια είναι κατά. Δύο, τρεις είναι υπέρ, κατά της τροπολογίας αυτής. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. 08 12 τοπολογίες 53, 66, 42, 49 και 79, 74. Η συγγήτρια είναι κατά και των τριών υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, 7 κατά. Και μία αποχή. 42, 50, 79, 75 και 53, 67 τροπολογίες. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 05-03-01-01. Τροπολογία 63-34. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ψήφι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 05-03-02-06. Τροπολογία 40-53. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ψήφι κατά. Θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σκοτάει κλού. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. 19 κατά, 12 υπέρ, 4 εποχές. Γραμμή 05030244, τροπολογία 8050. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Qui est Κατά. Ηλεκτρονικά και εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ 23 κατά 2 αποχές. 05-03-02-52 γραμμή. Τροπολογία 40-38. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. Γραμμή 05-04-05 01. 83-33 Ησίτα Η συγγύτα είναι κατά. Υπέρ. Ευχαριστώ. Ψήφι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 05-04-60-01. Η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Merci, baissez les mains, avis contraire. Είναι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11.06.60. 68-90. Υπέρ εισηγητρία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42-22. Αυτή έχει καταπέσει. Γιατί η 68-90 εγκρίθηκε. και θα τελειώσουμε τώρα με το δεύτερο κεφάλαιο. À la rubrique 3. Τελειώσαμε το 2 και πάμε στο 3. Τώρα έχουμε εδώ μια υπομάδα τροπολογιών, ώστε ε, να καλυφθούν κάποιες εγγραφές στον προπορισμό που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε εδώ στον πίνακα βαθμών 5 τις λεπτομέρειες. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ με ανατασή Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μια δεύτερη πομάδα τροπολογιών για να εγγραφούν κάποιες πιστώσεις πέραν των όσων είχε προτείνει η Επιτροπή. Έχετε τις λεπτομέρειε στον πίνακα 6. Ποιοι είναι υπέρ των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. 6 κατά. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται είναι τροπολογίες. Τώρα έχουμε 16.02.04 τροπολογία βαριθμών 2. Είναι κατά η εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Χωριστά. Μόνο αυτή. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 20, 16. 16.03.02.05 Ποιοι είναι υπέρ Κατά Αποχές την τροπολογία. 16.03.04 τροπολογία 1020. Είναι κατά. Η εισηγήτρια ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία εποχή. 03, 16.03.01 Είναι κατά εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 216. Υπέρ εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 17.03.52. 41-30. Με κατάσταση. Ποιοι είναι υπέρ. Δύο υπέρ. Κατά. απορριπτωτα 17 Απορρίπτονται. 17-04-04. Κατά εισηγητρία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18-02-01-01 Η 42-32 Υπέρ η Σεγγίτρια Ποιοι είναι υπέρ Ποιοι είναι κατά Απορρίπτεται ε, Για το ίδιο κονδύλι 7-40 Ποιοι είναι υπέρ 7-40 Ένας υπέρ. Τρεις. Ποιοι είναι κατά. Δεν έχουμε εποχές. Και απορρίπτεται. 18-02-01-02. Η 741. Είναι κατά η συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Καμία εποχή. Απορρίπτεται. 998. Κατά εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Με τρεις αποχές απορρίπτονται. Το ίδιο κονδύλι. Ε, για το 4164. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. 18.02.01.03 για 742. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18.03.01.01 για την 996 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 411 κατά εισηγήτρια ποιοι είναι υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 739 κατά σίδρα ποιοι είναι υπέρ Έχετε δίκιο γιατί εγκρίθηκε η 411 και οι υπόλοιπε καταπίπτουν. But comme le, comme le 996 n'a pas été adopté, μια που δεν εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή θα πρέπει να πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. 739. 739 είναι κατά εισηγήτρια. Vérification des votes sur le 411. Yeah. Για το 411 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Είναι κατά εισηγήτρια. Ψηφίζουμε. Vous avez voté Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε το 411 και εγκρίνεται. Τριάντα έξι. Αφού γίνεται το 411, τότε το 739 καταπίπτει. Και το 4162 επίσης. 18.03.01.02 το 997 κατά εισηγήτρια υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το 997 πέρας απορρίπτεται 13-23 737 κατά εισηγητρία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41-63. Κατά εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αμφιβάλλεται. Όχι. Προχωρούμε. στο 412. Κατά η συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, γιατί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Για το 412. Πέρασε. Κρίνεται. 19-17 και μια εποχη αποχή 18-03-03 ή 776 Εισηγήτρια πίνει υπέρ κατά αποχές ανέχομαι απορρίπτεται 1001 Χίλιαν, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40-35. Υπέρ. Η Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. τρεις κατά, χωρίς αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη. Κατάρρηση γήτρια. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δύο αποχές απορρίπτεται 33.02.01 η 999 κατά εισηγήτρια υπέρ κατά απορρίπτεται 752. Κατά εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 381. Υπέρ. Η εισηγήτρια υπέρ. Κατά. 3 κατά δύο εποχές. Η τροπολογία εγκρίνεται και τώρα πάμε στο 330202. Το 732. Κατά η εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. Χίλια. Κατά εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές καμία απορρίπτεται 738 ταυτόσημη ε, ποιοι είναι υπέρ είναι κατά ποιοι είναι κατά αποχές απορρίπτεται 41-65 Κατά. Η εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 406 υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις κατά Τώρα, οι οι οποίε αφορούν κάποια σχόλια ή παρατηρήσει για το 16.02.01. Η τροπολογία 69.05. Υπέρ ή εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. 4.009. Υπέρ, η εισήγητρια. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16.03.01 για το 52.23. Πέρ, εισήγητρια. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές κρίνεται. η 80-60 υπέρ συγκίτρια ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές τρεις απορρίπτεται η τροπολογία 170401 4136 είναι κατά εισηγητρία ποιοι είναι υπέρ είναι κατά αποχές και απορρίπτωση Nous en venons à la ligne 1704. 17-04-02. 42-46 χωριστή ψηφορία. Πρώτα-πρώτα. Μιλούμε για τους παράγοντες που απειλούν την γεωργία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. 5 απορρίπτεται. Αυτό το τμήμα το οποίο σας ανέφερα και τώρα. Μετά που αφορά την αρρωγή προς τους ε, καλλιγητές υπέρ η συγγήτρια, ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας, ποιοι είναι κατά, αποχές, τρεις αποχές, απορρίπτεται. 79-71. Κατά εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 62-55. Και εδώ έχουμε χωριστέ τρεις ψηφοφορίες για αυτή την τροπολογία. Πρώτα από τα παράνομη μετανάστευση είναι υπέρ η εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται γιατί έχουμε ισοψηφία. Ακόμα μια ψηφορία όσον αφορά το δεύτερο τμήμα και που λέμε για την προοπτική των δύο φύλων. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Αυτό το τμήμα εγκρίνεται. 19-14. Με δύο εποχές. Και τώρα πάμε στο τρίτο, τρίτο τμήμα που αφορά μια προσέγγιση η οποία είναι ευαίσθητη στην ισότητα των φύλων. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με 34 εκτές τροπολογίες και τώρα πάμε στο 83-43. Δεν έχουμε ψηφίσει. Ε, αλλά καλύπτεται το 62-55 και πάμε στο επόμενο. 62-16 υπέρ εισηγήτρια. 62-16 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα, ηλεκτρονικά. Πέρας. 19-15 εγκρίνεται. 62-18. Υπέρ εισηγητρία. ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται 21, 29, 3. Επόμενο κονδύλιο με την τρεις διχορτές ψηφορίες για την 62-19. Πρώτα-πρώτα, παράνομη μετανάστευση. Υπέρ εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Ναι, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκαεννέα, δεκαεπτά. Οπτική γωνία, σώτος φύλλων, ψηφίζουμε. Αυτό το τμήμα εγκρίνεται. 19-16. Τρίτο τμήμα της, της ε, τροπολογίας, παραμετανάστευση, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ανθρωπιών όντων, είναι υπέρ εισηγήτρια. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 30 υπέρ 3 κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο επομένω τη τροπολογία αυτή εγκρίνεται. 33.02.01. Ψηφίζουμε χωριστά τρία τμήματα. Δάφνη πρώτα-πρώτα. Υπέρ εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αυτό το τμήμα της τροπολογίας, το, το δεύτερο. Στατιστικά τα οποία έχουν περισυλλεγεί και έχουν ε, ε, αποτελέσει ένα σύνολο ανάλογα με το ποιο φύλλο αφορούν. Υπέρ, κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Το τρίτο τμήμα της τροπολογίας, αυτό η προσέγγιση από οπτικής γωνίας των ισότητων των δύο φύλων, υπέρ, Ευχαριστώ. Κατά. Να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. 17-14 χωρίς αποχές συγκρίνεται. 33 πρώτον στατιστικά ανά φύλλο υπέρ ηλεκτρονικά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά είναι 31-3. Και όσον αφορά την πρικοδότηση του προπολογισμού του, των πολιτικών για ισότητα των φύλων, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. 17, 14, 3 αποχές. Εγκρίνεται. 83-42 καλύπτεται από αυτήν που, που ενεκρίθη. 61-67 υπέρ εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. ηλεκτρονικά. Πέρας. Η Εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώσαμε το τμήμα 3. Αν μπορούσαμε να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά λόγω της ε, εξαιρετικής προπαρασκευής από την εισηγήτρια, μπορέσαμε να προχωρήσουμε κι άλλο. Οπότε θα μπορούσαμε να διεξαγάγουμε και την ψηφορία, αν συμφωνείτε, για τα ειδικά μέσα εργαλεία. Συμφωνείτε να συνεχίσουμε. Συμφωνείτε να συνεχίσουμε την ψηφοφορία για να μπορέσουμε να έχουμε λιγότερα να εξαγάγουμε αύριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 1α πρέπει να ψηφίσουμε. Είμαστε έτοιμοι για το 1α. Εάν θέλουν ε, οι άλλες πολιτικές ομάδες να συνεχίσουμε. Εάν όχι, δεν είναι έτοιμες οι άλλες πολιτικές ομάδες, τότε αύριο. Ε, από εσάς Δεν σας είδα. Κύριος Ντεπρέ. Για αύριο. Αύριο θέλουμε. Και ευχαριστώ για την ε, πρόσφορα του κύριου Φεραντές να αναβάλουμε. Τι λέτε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν να συνεχίσουμε αύριο. Αλλά μην φύγετε. Να σας ευχαριστήσω γιατί προχωρήσαμε Οπότε διακόπτουμε και θα συνεχίσουμε αύριο σε 9.30 ώρα. 9, 9 διορθώνει ο πρόεδρος. 9, 9 η ώρα. 9.